Επομένως, έχει επικυρωθεί και από την Ολομέλεια ο έλεγχος της εντολής. Η Επιτροπή Συνταγματικών Θεμάτων προτείνει βάσει του άρθρου 117 παράγραφος 3 να δοθεί γραπτή απάντηση σε μία σειρά κειμένων. Τα κείμενα αυτά είναι στη διάθεσή σας. Οποιαδήποτε ένσταση θα πρέπει να διατυπωθεί μέχρι αύριο το πρωί από μία πολιτική ομάδα ή τουλάχιστον 40 βουλευτές, όπως αναφέρεται στο άρθρο 211. Σε σχέση λοιπόν με τα κείμενα